Καθίστε παρακαλώ. Η, συνεδρίαση και η ακρόαση ξεκινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον προτινόμενο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για την ακρόαση αυτή από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά το τέλος εβδομάδας ε, θα έχουμε ακρόαση και με την ε, προτινόμενη Επίτροπο Γιώροβα για θέματα δικαιοσύνης και με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Σήμερα όμως θα έχουμε ακρόαση με τον προτινόμενο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τα θέματα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων είναι ο πρώτος επίτροπος που έχει στο χαρτοφυλάκιό του τη μετανάστευση. Και νομίζω όλοι έχουμε επίγνωση της τεράστιας σημασίας αυτού του θέματος. Με βάση το παράρτημα 16 του εσωτερικού κανονισμού που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τον προτινόμενο, τους προτινόμενους επιτρόπους με βάση τις γενικές τους ικανότητες, την ευρωπαϊκή τους αφοσίωση και την προσωπική του ανεξαρτησία θα εκτιμήσει και θα αξιολογήσει τη γνώση των χαρτοφυλακίων τους και τα επικοινωνιακά τους προσόντα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο στους προτινόμενους επιτρόπους με δύο κοινέ ερωτήσεις που έχουν συντάξει οι πρόεδροι στη διάσκεψη των πρόεδρων και τρεις ειδικέ ερωτήσεις της δικής μας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ο προτινόμενος επίτροπο απάντησε γραπτό στο ερωτηματολόγιο αυτό και σας έχουμε μοιράσει μεταφρασμένες απαντήσεις. Η δομή της συζήτησης θα έχει ως εξής. Ο προτινόμενος επίτροπος θα κάνει μια εισαγωγική αρχική παρουσίαση το πολύ 15 λεπτών. Μετά την εισαγωγή θα έχουμε χρόνο για υποβολή 45 ερωτήσεων από τα μέλη και απαντήσεις από τον Επίτροπο. Τρία λεπτά για κάθε ερωταπάντηση. Ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων θα θέσουν ερωτήσει εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Κατά το τέλο τη ακρόαση, ο προτινόμενο επίτροπο θα έχει ένα επιπλέον πεντάλεπτο για τα τελικά του σχόλια. Λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου. Γιατί αν δεν σεβαστούμε το χρόνο μα, δεν θα περισσέψει χρόνο για να μιλήσουν όλοι και θα χρειαστεί να, θα χρειαστεί να διακόπτω ε, τους ομιλητές. Έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες, οπότε ο καθένας μπορεί να μιλά και να ακούει τη μητρική του γλώσσα. Δεδομένου ότι έχουμε διερμηνία, σας θερμοπαρακαλώ να μιλάτε αργά και καθαρά. Επίσης γίνεται απευθείας αναμετάδοση της ακρόασης από το ε, διαδίκτυο και μπορείτε αργότερα να δείτε και μαγνητοσκόπηση της ακρόασης. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν θα δώσω το λόγο στον προτινόμενο μας επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο για την παρουσίασή του. Κύριε Αβραμόπουλα, έχετε το λόγο για 15 λεπτά.